Καλημέρα σας. Βλέπω ότι είμαστε πολύ μεταξύ μας. Άρχεται η συνεδρίαση. Υπάρχει μία ανακοίνωση. Η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα ξεκινήσει τις ε, διαθεσμικές διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 69C, παράγραφος 1 του κανονισμού. Τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας, δυνάμει του κανόνα του άρθρου 69 69Γ, παράγραφος 2, μέλη ή πολιτικές ομάδες που φτάνουν σε ένα συγκεκριμένο κατόφλι μπορεί να ζητήσουν μέχρι αύριο, Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στις 12 τη νύχτα, να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις δυνάμει ψηφοφορίας. Εάν δεν υπάρξει τέτοιο αίτημα από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορούν να αρχίσουν, μπορεί η Επιτροπή Λίμπε να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις. Τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Γκαρντίνη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σήμερα νομίζω ότι θα γράψουμε μία πολύ ωραία σελίδα της ευρωπαϊκής ιστορίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ε, τους εμπλεκόμενους αρχίζοντας από τους και όδης, αλλά και ολόκληρο το Κοινοβούλιο, το οποίο με την ευελιξία του και την δυνατότητα να ε, διαβλέψει την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού πολιτικής, πολιτικής προστασίας να κατάφερε να μπορέσει να ξεπεράσει ορισμένες αμφιβολίες κρατών μελών, έτσι ώστε η πολιτική προστασία να μην θεωρηθεί παρεμβατισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι πολίτες θέλουν την πολιτική προστασία και θέλουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλάι τους τη στιγμή που οι τοπικές και περιφερειακές αρχές δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έκτακτες καταστάσεις. Είδαμε τι ε, έγινε με τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Πορτογαλία και την Ελλάδα, όπου χάθηκαν πολλές ε, ζωές πέρα από τις ε, οικονομικές ζημίες. Γι' αυτό χρειάζεται αυτός ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, γιατί δεν μπορεί να γίνει αντιμετώπιση σε τοπικό ή κρατικό επίπεδο πάντα. Ένα χρόνο μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τη σπουδή με την οποία ε, αντιμετώπισε το θέμα ο Επίτροπος Στυλιανίδης, έχουμε το RESC-EU. Το RESC-EU είναι ένα νέο μέσον που απαρτίζεται από επιπρόσθετους πόρους σε σχέση με τους προϋπάρχοντες και που είναι των κρατών μελών. Γιατί το RESC-EU θέλει ακριβώς να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα εκεί όπου χρειάζεται, μέσα στα πλαίσια και της πρόληψης και της προετοιμασίας έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις φυσικές καταστροφές είτε όταν πρόκειται για ατυχήματα τα οποία προκύπτουν από την χρήση χημικών ουσιών, πυρηνικά ατυχήματα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι οι πυρκαγιές είναι υπεύθυνες για το 20% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτόν τον ενισχυμένο μηχανισμό. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ως Ιταλίδα να σας πενθυμίζω τον Τζουζέπε Τζαμπερλέτη που είναι ο θεματοφύλακας της πολιτικής προστασίας και θα ήθελα να του αφιερώσω αυτή την ημέρα και αυτή την εργασία, κύριε Επίτροπε, γιατί πέρα από ένα είδος εράσμου στο οποίο θεσμοθετήθηκε και που αποτελεί ε, έναν κοινό παρονομαστή όλων, υπάρχει και ο μηχανισμός αναγνώρισης για εκείνους ε, οι οποίοι διακρίθηκαν στο τομέα της πολιτικής προστασίας. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, θυμίσω την ύπαρξη αυτού του μεγάλου ανθρώπου και νομίζω ότι σήμερα μας στέλνει και εκείνος ένα μεγάλο χαμόγελο για αυτή την εργασία. Ευχαριστώ κυρία Καρδίνη. Ναι, και εγώ θα ήθελα να πω ότι γνωρίσαμε πολύ καλά τον κύριο Τζαμπερλέτη, ο κύριο Ζόφκο από την Επιτροπή, η κυρία Ζόφκο, από την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια, να συγχαρώ την κυρία καρδίνη διότι έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο θέμα της έκθεσής μας, την πολιτική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Επίτροπο κύριο Στυγιαννίδη. Ήμουν εισηγήτρια προς γνωμοδότηση από την Επιτροπή Ανάπτυξης και θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη να, ενισχυθεί, να ενισχυθούν και οι εθνικές ικανότητες πολιτικής προστασίας και οι διεθνείς συνεργασίες, επιτρέποντας τους μηχανισμούς στις διάφορες χώρες ε, μέλη να λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Το νέο εργαλείο πρέπει να έχει στόχο την πρόληψη κινδύνων. Είχαμε πολλές πυρκαγιές ε, δασών τα τελευταία χρόνια, ιδίως στην Νότια Ευρώπη και χρειάζεται από πλευράς μας να υπάρξει μια ισχυρή αντίδραση. Θα ήθελα να ζητήσω οι χώρες εκείνες που δεν μπορούν να μετάσχουν πλήρως, να λάβουν κάποια χρηματοδότηση για τη μεταφορά, 50% ενδεχομένως. Αυτό για την Κροατία, για παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό. Η Κροατία χρειάζεται μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων για όλα τα μέτρα ε, πολιτικής προστασίας. Επίσης, ο μηχανισμός Rescue θα πρέπει να επιτρέπει πάντα στα κράτη-μέλη να ελέγχουν την ανάπτυξη των δυνάμεων στο κράτος, στα κράτη-μέλη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για τον μηχανισμό αυτό που θα επιτρέψει στους πολίτες της Ένωσης να μην αισθάνονται απομονωμένοι πλέον. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στυλιανίδης, ο Επίτροπος, έχει το λόγο και εγώ τον ευχαριστώ για την παρουσία του στην Ολομέλεια σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι, μίλησα στη, στο Κοινοβούλιο πριν από ένα χρόνο περίπου, παρουσιάζοντας την πρότασή μας για την ενίσχυση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, μετά από ένα χρόνο, το Κοινοβούλιο ψηφίζει την πλέον φιλόδοξη, το πλέον φιλόδοξο σύστημα πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη που έχει υπάρξει ποτέ. Σήμερα το Κοινοβούλιο ψηφίζει κάτι που ήταν πολιτικά διανόητο πριν από λίγα χρόνια. Είμαστε φίλοι εδώ τώρα και θα σας τα πω με ειλικρίνεια. Ήταν πολύ απαιτητική δουλειά, πολύ δύσκολη δουλειά να πείσω τα κράτη να δεχθούν αυτή την προσέγγιση. Εν τέλει όμως καταφέραμε και υλοποιήσαμε αυτό τον πολύ φιλόδοξο κοινό στόχο. Σήμερα λοιπόν είμαι πραγματικά περήφανος που είμαι Ευρωπαίος. Θέλω πρώτα πρώτα να, ευχάσω, να ευχαριστήσω ειλικρινά την εισηγήτρια κυρία Γκαρντίνη για την ηγετική θέση που έλαβε στην, στο να προωθήσει το σημείο αυτό στο Κοινοβούλιο και όλους τους συναδέλφους την κυρία Ζόφκο τον κύριο Ενάντες και όλους τους σκιώδεις εισηγητές από τις πολιτικές ομάδες τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ολόκληρο που υποστήριξαν με πάθος αυτό το ρηξικέλευθο μέτρο. Συνάδελφοι, με την πολιτική σας υποστήριξη το Rescue θα είναι εκεί παρόν στις επόμενες δασοπυρκαγιές. Και χάρη στην δική σας αφοσίωση στον κοινό μας στόχο, για την προστασία των πολιτών μας, για την διάσωση ανθρώπινων ζωών και των σπιτιών τους. Πραγματικά ζητήσατε εγγύηση για καλύτερη και άμεση διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στις καταστροφές. Και σήμερα μπορώ να σας πω το εξή. Συνεργαζόμαστε στενά με τα κρατη για να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό την μεταβατική φάση του rescue, όπως το λέμε, ούτως ώστε να μπορούν να υπάρξουν ικανότητες ε, ανταπόκρισης της κρίσης για την Ευρώπη ήδη φέτος. Η ενημέρωση και οι πληροφορίε που παίρνω από τα κράτη-μέλη μέχρι τώρα είναι πολύ θετικέ και ευχαριστώ και εγώ τα κράτη-μέλη σήμερα για την θετική τους προσέγγιση. Βέβαια, μην βαφκαριζόμαστε δεν θα σταματήσουν οι φυσικέ καταστροφέ. Αντίθετα θα γίνονται συχνότερε και πιο έντονε λόγω τη αλλαγή του κλίματο. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το νέο αυτό φαινόμενο τη αλλαγή του κλίματο όσο καλύτερα μπορούμε. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με το Rescue είναι να εξοπλίσουμε καλύτερα και του εαυτού μα και τα κρατημέλη για να αντιμετωπίσουν καλύτερα τι καταστροφέ από την αλλαγή του κλίματος. Η νέα αυτή νομοθεσία κύριε και κύριοι δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη και την προπαρασκευή. Το Κοινοβούλιο κατέστησε σαφές ότι τούτο ήταν προτεραιότητα για εσά και κάναμε ό,τι μπορούμε για να θεσπίσουμε ένα σύστημα που παρέχει περισσότερη υποστήριξη στα κράτη για την ανταλλαγή πληροφοριών και για να διδαχθεί το ένα από το άλλο. Συνάδελφοι, σήμερα με μετριοφροσύνη μπορώ να πω ότι χαράσουμε το ξεκίνημα μιας νέας εποχής πολιτικής προστασίας στην Ευρώπη. Μιλάμε για μια Ευρώπη που προστατεύει. Αυτό το οφείλουμε, όπως είπα, στους πολίτες μας. Κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε περήφανοι λόγω του επιτεύγματος αυτού και θέλω εκ νέου να σας ευχαριστήσω για την αφοσίωση και την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την Επιτροπή Προϋπολογισμών ο κύριος Φερνάντες ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρώπη που προστατεύει αποτελεί μία αναγκαιότητα. Η προστασία της ανθρώπινας ζωής θα πρέπει να είναι το βασικό μας μέλημα. Το 2017 στην Πορτογαλία ζήσαμε μία μεγάλη τραγωδία. Πάνω από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί. Ο νέος αυτός μηχανισμός δείχνει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι ο επιμερισμός των ευθυνών, ιδιαίτερα όσον αφορά την πολιτική προστασία. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να στοιχηματίζουμε στην πολιτική προστασία και η προστασία είναι το βασικό μας μέλημα. Επίσης, πολλοί υπουργοί οικονομικών δεν δέχτηκαν αυτή την συμφωνία και τι έκαναν, διαπραγματευτήκαν ένα ποσό 100.000 ευρώ, δηλαδή ένα μελιτέο ποσό για το 2019. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την δέσμευση του κυρίου Στυλιανίδη και της κυρίας Γκαρντίνη, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία συμφωνία που δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή ε, ένωση σώζει ζωές και αυτό πραγματικά αξίζει. Η κυρία Μίλναρ δεν είναι παρούσα, άρα περνάμε στις πολιτικές ομάδες. Για το ΕΛΚ ο κύριος Γκαμπής για 1,5 λεπτό. Θα ήθελα όλοι να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ η Ευρώπη δημιουργείται μέσω της αλληλεγγύης και της αδελφοσύνης μεταξύ των λαών της. Αυτή είναι μια αρχή που σήμερα περισσότερο παραποτέ πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ στο ημικύκλο στο Στρασβούργο. Η αλληλεγγύη μεταξύ των Ευρωπαίων δημιουργείται από κάτω προς τα πάνω και με βάση αυτή την πιο βασική ανάγκη που είναι η αντιμετώπιση των απροβλέπτων ε, θεομηνίων όπως είδαμε στις τεράστιες πυρκαγιές στην ε, Πορτογαλία και την Γαλλική του 2017. Όμω πρέπει να είμαστε και έντιμοι μεταξύ μας. Κάτι λείπει όταν η Ευρώπη δεν είναι η πρώτη που να ανταποκρίνεται όταν υπάρχει μια τέτοια θεομηνία. Γι' αυτό θεωρώ ότι η δημιουργία του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας είναι ένα καλό εργαλείο που μπορεί να συνδυαστεί με την πρόταση για αυτό το σώμα Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Και έτσι θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για την Ένωση, για να δείξουμε ότι μέσω της ενότητας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, τη συνάδελφο Γκαρντίνη, για την εργασία της για το θέμα αυτό, για το καλό αποτέλεσμα που επέτυχε και για τη λειτουργικότητα και την άμεση επίπτωση που θα έχει αυτός ο μηχανισμός στο μέλλον στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Ανδρουλάκης. Ε, παρακαλώ, Νίκο, δυόμιση λεπτά. Τελευταία χρόνια, σε πολλούς από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι θεσμοί μοιάζουν απόμακροι, ακόμα και εχθρικοί όμως στην περίπτωσή μας η αγωνία τους για καλύτερη προστασία από φυσικές καταστροφές αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας ένα πραγματικό εργαλείο αλληλεγγύης δημιουργώντας το resceu. σήμερα η ανθρωπιά και η στήριξη των λιγότερο δυνατών και η περιβαλλοντολογική ηθική είναι νικητές. η αφορμή για τη συγκεκριμένη πρόταση ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην πορτογαλία. κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις μια νέα τραγωδία θα έπληκε την ευρώπη. αυτή τη φορά στο μάτι λίγο έξω από την αθήνα με πάνω από 100 νεκρούς. αυτά τα γεγονότα κατέσαν σαφές σε όλους ότι πρέπει να προσφέρουμε μια ουσιαστική απάντηση στις ανησυχίες των πολιτών σε αυξανόμενε φυσικέ καταστροφέ λόγω κλιματική αλλαγή ή ανεπαρκή προετοιμασία από τι εθνικέ αρχέ δεν μένουμε παρατηρητέ αλλά δίνουμε μια ισχυρή απάντηση. όλοι μαζί με περισσότερη οργάνωση μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα από ότι ο καθένα μόνο του. ο δρόμο τη πολιτική ενοποίηση είναι μακρύ και γεμάτο εμπόδια που βάζουν οι θειασότε μια ευρώπη όπου η αλληλεγγύη δεν είναι αυτό σκοπό αλλά μέσο με κόστο που δεν θέλουν να αναλάβουν ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. δημιουργούμε το resceu μια ευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων όπως πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα τα οποία θα αγοραστούν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 80 έως 90% των συνολικών εξόδων διασφαλίζοντας ότι καμία χώρα δεν θα μείνει ξανά αβοήθητη. παράλληλα για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έως 75% για τη συντήρηση των εθνικών μέσων. η βοήθεια αυτή σε χώρες όπως η ελλάδα που η αδυναμία επισκευής λόγω της οικονομικής κρίσης έχει περιορίσει πάρα πολύ τη δράση των εθνικών μέσων είναι απαραίτητη. τέλος ενισχύουμε την πρόληψη διατηρώντας ανώθευτα τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης. απορρίψαμε την πρόταση του συμβουλίου που προέβλεπε την εισαγωγή ποινών για τι χώρε που ζητούν συχνά την ενεργοποίηση του μηχανισμού. αντιθέτω δίνουμε τη δύναμη στην επιτροπή να εξετάσει τα μέτρα πρόληψη του συγκεκριμένου κράτου και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνει να υπάρχουν συστάσει για βελτίωση ή ενίσχυση των εθνικών σχεδίων προστασία. όλοι οι ευρωπαίοι πολίτε ανεξάρτητα του κράτου μέλου που κατοικούν πρέπει να νιώθουν ασφαλεί και να ξέρουν ότι η ένωση μπορεί να του βοηθήσει με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση μια έκτακτης ανάγκης. Για την, συντηρητικού συντηρητικού ο κύριος Γκέρικε. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Από πλευρά ε, των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γκαρντίνη η οποία ασχολήθηκε με αυτή τη διοργανική συμφωνία που ανταποκρίνεται σε όλα τα ε, αιτήματά μας και συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Έτσι θα έχουμε ιδιαίτερε υπηρεσίε διάσωση που θα βοηθούν τα κράτη-μέλη αν θα <coughs> συμπεραστεί από τα γεγονότα οι δικέ του υπηρεσίε. Όπω ιδιαίτερα κατά τι ε, δασοπυρκαγιέ ε, το περασμένο καλοκαίρι. Ελπίζουμε μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε ειδικά ε, πυροσβεστικά αεροπλάνα για να καταπολεμήσουμε τι πυρκαγιέ που κατά πάσα πιθανότητα και πάλι θα προκύψουν. Θεωρώ ότι πετύχαμε λοιπόν τη συνεργασία Κάτι που σπάνια έχουμε επιτύχει στο μέλλον, ούτως ώστε η αντιμετώπιση των καταστροφών να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές. Και έτσι νομίζω ότι είμαστε πρωτοπόροι όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παγκοσμίω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γιάτενμα και 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και την κυρία Γκαρντίνη. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι τελικά η κύρια ευθύνη για την πολιτική προστασία εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια των κρατών μελών. Οι ενωσιακοί πόροι θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως σύστατη προσφυγή. Κανένα κράτος μέλος ούτως ή άλλως όμως δεν θα πρέπει να δώσει ως υπεργολαβία την πολιτική προστασία σε άλλες χώρες αυτό θα ήταν και επικίνδυνο και ανεύθυνο. Ξέρουμε ότι όταν ε, υπάρχει μια θεομηνία πρέπει κανείς να δράσει ε, τάχιστα διότι τα πρώτα λεπτά, οι πρώτες ώρες ε, είναι πιο σημαντικές για την αντιμετώπιση της. Αν περιμένουμε να έρθουν από αλλού οι αρμόδιοι της πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τότε οι επιπτώσεις θα είναι πραγματικά τραγικές. Η πρόληψη φυσικά είναι πάντα καλύτερη από την αντιμετώπιση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ έχει ρόλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίξει τα κράτη-μέλη και για την πρόληψη και για την αντίδραση βεβαίως. Όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν και βεβαίω και η διαλειτουργικότητα ε, του εξοπλισμού είναι αναγκαία. Αλλά το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει αυτό και μόνο να έχει την αρμοδιότητα για να έχει διαθέσιμο το κατάλληλο εξοπλισμό εάν υπάρξει πρόβλημα αλλά και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι βεβαίω και αυτή πολύ σημαντική. Αναφέρθηκαν οι δασοπυρκαγιέ. Και εδώ η πρόληψη είναι ιδιαίτερα σημαντική για να αποφεύγονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παπαδημούλη για την ΚΟΕ, ένα λεπτό. Είναι μία από τις λίγες θετικές ειδήσει που παράγουμε ως Ευρωπαϊκή θεσμοί το τελευταίο διάστημα και αυτό το οφείλουμε στην πίεση του Ευρωκοινοβουλίου, στις θετικές προσπάθειες του Επιτρόπου Στυλιανίδη και στη συνεργασία Ευρωκοινοβουλίου Κομισιών που έκαμψαν τις αντιρρήσεις ορισμένων κρατών μελών. Γιατί ήρθαν και τα γεγονότα να βοηθήσουν. Τα τραγικά γεγονότα. Οι μεγάλες πυρκαγιές στην Πορτογαλία. Φωνικές οι πυρκαγιές στην πατρίδα μου την Ελλάδα και οι πλημμύρες φωνικές, οι σεισμοί στην Ιταλία, με νεκρούς επίσης, αλλά και οι μεγάλες πυρκαγιές στη Σουηδία που έκαναν και τους βόρειους τα βόρεια κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν απειλεί μόνο τον Νότο και ότι χρειαζόμαστε μια επικουρική δύναμη ευρωπαϊκή να ενισχύει τις προσπάθειες των κρατών μελών. Και έπαψε αυτή η ευρωτσιγκουνιά. Και έχουμε περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Και η τελική πρόταση είναι βελτιωμένη χάρη στην επιμονή του Ευρωκοινοβουλίου και κινείται σε θετική κατεύθυνση. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει και μια ευρύτερη στήριξη μέσα στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τις απόψεις των πολιτικών ομάδων. Κάποιοι αγορητές ή, ατομικά. Ο κύριος Μάντελ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Ο χειμώνας στην Αυστρία απέδειξε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης, οι εθελοντές, οι πυροσβέστες και οι άλλες ε, δυνάμεις για την αντιμετώπιση είναι θαυμάσιες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να έχουμε την ε, ε, δυνατότητα να μην χρειαζόμαστε βοήθεια εκ των έξω όταν προκύψουν απρόβλεπτες καταστροφές οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Είναι σωστό λοιπόν που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα μηχανισμό αντιμετώπισης καταστροφών. Και συμμερίζουμε αυτό που είπαν ήδη ε, επανειλημμένα οι συνάδελφοι, ότι εμείς ως Κοινοβούλιο βελτιώσαμε ιδιαίτερα την έκθεση. Είναι λιγότερο συγκεντρωτική, λιγότερο γραφειοκρατική και χαίρομαι που η Προεδρία του Συμβουλίου είναι τώρα στην ε, Αυστρία και αυτή θα ολοκληρώσει αυτή την επιτυχία. Και εμεί επίση μπορούμε να κρίνουμε το τελικό αποτέλεσμα. Διότι η αρχική πρόταση τη Κομισιόν που προέβλεπε κέντρα ε, ελέγχου και παροχή εντολών. Καταλήγουμε τώρα σε ένα πακέτο που στηρίζει περισσότερο την συνεργασία και πρώτα απ' όλα την ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών μηχανισμών ασφαλείας. Αυτό είναι το παράδειγμα της Αυστρίας και έπαιξε ένα ρόλο νομίζω στη διαμόρφωση της τελικής πρότασης. Και βεβαίως θα πρέπει κυρίως να βασιζόμαστε στις ε, δικές μας δυνάμεις. Σήμερα κάναμε ένα σημαντικό βήμα για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας έτσι ώστε να μπορέσουμε συντονισμένα να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη. Οι καταστροφές ήταν συντριπτικές για ολόκληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Γι' αυτό χρειάζεται αυτός ο πολιτισμός πολιτικής προστασίας παντού και όχι μόνο στο Νότο και γι' αυτό χρειάζονται και η κατάλληλη πόλη. Πιστεύω ότι η δημιουργία αυτού του αποθεματικού ΡΕΣΚΙΓΙΟΥ είναι ύψη της σημασίας και η συζήτηση και η έκθεση μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε αυτή την προσπάθεια, να συγχαρούμε την εισηγήτρια και ελπίζουμε να έχουμε και την στήριξη των κρατών μελών για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε όλους τους κινδύνους. Ε, κύριε Επίτροπε, όμως αυτή η πολιτική ε, δεν μπορεί να αναβληθεί για το μέλλον. Θα πρέπει να υπερβούμε τους γραφειοκρατικούς ε, μηχανισμούς και αυτό μέσα στα πλαίσια και του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 21-27. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το χρονοδιάγραμμα της πρότασης νομοθετικού περιεχομένου. Εάν λοιπόν δημοσιευτεί σήμερα, ήδη θα ήταν αργά. Θα πρέπει να αποτρέψουμε τις φυσικές καταστροφές. Χρειάζονται οι πολίτες το Rescue ήδη. Φερέιρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία των κρατών μελών, ιδιαίτερα για τις καταστροφές μεγάλων διαστάσεων. Χρειάζεται συντονισμός προσπαθειών και επιμερισμός ευθυνών. Η Ευρώπη δεν έχει κάνει ό,τι μπορούσε σε αυτό το τομέα. Η κατάσταση το 2017 στην Πορτογαλία ε, καταδεικνύει την κατάσταση. Οι πυρκαγιές στην Πορτογαλία ήταν καταστροφικές. Και δυστυχώς θα υπάρξουν και περικοπές από όσο προβλέπεται, ακόμα και για την πρόληψη των καταστροφών. Δυστυχώς δυστυχώς οι καταστροφές πλήττουν χώρες που δεν έχουν τόσο σοβαρά μέσα στη διάθεσή τους για να τις αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν την εποπτεία αυτού του μηχανισμού. Διαφορετικά, αν υπάρχει αποκέντρωση, τότε ελοχεύουν κίνδυνοι και πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Ε, Καπεθόν Ρουίθ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αρχίζει να λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός που σημαίνει περισσότερη Ευρώπη, Ευρώπη αλληλεγγύης, ούτω ώστε να προλαμβάνουμε και να αντιμετωπίζουμε και να απαλύνουμε τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών. Αλλά τονίζω ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης που πρέπει να δώσει αποζημιώσεις για τις φυσικές καταστροφές. Είναι σημαντικό, όπως έχουμε ζητήσει, να συμπεριληφθεί και το περιβάλλον να ληφθεί η υπόψη η οικονομική ζημία από τις περιβαλλοντικές καταστροφές για να δίδονται αποζημιώσεις. Είναι σημαντικό οι περιφέρειες που θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτό το ε, ταμείο να υπολογίζονται με βάση το τοπικό ΑΕΠ και όχι το ΑΕΠ ολόκληρης της αλληλεγγύης. Έτσι μόνο θα αντιμετωπίσουμε τις ε, ε, καταστροφές που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Θέλω λοιπόν να κάνω μία έκκληση να βοηθήσει και αυτό το ταμείο Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μεταρρύθμιση του κανονισμού του. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μαριά, ένα λεπτό. Οι φυσικές καταστροφές δυστυχώς είναι στην ημερήσια διάταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω φυσικά των κλιματικών αλλαγών. Και είχαμε τεράστιες καταστροφές, είχαμε τις ε, φωνικές πλημμύρες στη μάνδρα της Αττικής, τις φωνικές πυρκαγιές στο Μάτι με 100 νεκρούς, πυρκαγιές επίσης φωνικές στην Πορτογαλία, σεισμούς με νεκρούς στην ε, Ιταλία. Όλα αυτά δείχνουν ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας αποφασιστικό που να ενσωματώνει στην πράξη την αρχή της αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι τα βήματα που γίνονται είναι σε μια θετική κατεύθυνση. Θα πρέπει να καταλάβουν τα κράτη-μέλη ότι δεν μπορούν να επιβάλλουν ποινές στις χώρες οι οποίες θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχανισμό διότι η αξιοποίηση αυτού του μηχανισμού προέρχεται δυστυχώς λόγω των φυσικών καταστροφών. θεωρώ ότι πρέπει να πάρουμε ακόμη πιο αποφασιστικά μέτρα να στηρίξουμε τις χώρες που υφίστανται τις φυσικές καταστροφές και αυτές κυρίως είναι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου. ευχαριστώ. Η κυρία ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η σημερινή συζήτηση καταδεικνύει άλλη μια φορά σαφέστατα ότι η προστασία από τις καταστροφές και αντιμετώπιση αφορά πολλά θέματα, τη χωροταξία, την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση, πρώτα απ' όλα βεβαίως η πρόληψη. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστροφές. Χρειαζόμαστε καλή παρακολούθηση και νομίζω ότι η συζήτηση και η απόφαση που ελπίζω θα ληφθεί για αυτό το μηχανισμό θα συμβάλλει ιδιαίτερα ούτω ώστε στο μέλλον να μπορούμε να πούμε στους ε, συμπολίτες μας ότι αν υπάρξουν θεομηνίες η Ευρώπη βοηθάει όλοι μαζί. Δεν αφήνουμε μόνο τους, ε, τα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές. Όχι. Εμείς, εάν υπάρξει σοβαρή περίπτωση, η Ευρώπη είναι στο πλευρό τους. Με οικονομικούς πόρους, με τεχνικό εξοπλισμό, με τεχνογνωσία, για να βοηθήσει να απαλληλθούν οι συνέπειες των καταστροφών ή ακόμη και οι συνέπειε των καταστροφών που έχουν προκαλέσει τα άτομα, ούτως ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις όσο ταχύτερα γίνεται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόπε, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το θέμα που μας απασχολεί είναι πολύ σημαντικό σε κάποιες περιπτώσεις ε, το κράτος μέλος, ένα κράτος μέλος μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Για παράδειγμα, ο πυρηνικό σταθμό του Αστράβο στη Λευκορωσία. Ξέρουμε ότι η κατασκευή αυτού του πυρηνικού σταθμού έγινε κατά παράβαση των διεθνών προτύπων ε, για το ζήτημα αυτό. Τούτο γίνεται 20 χιλιόμετρα από τα, από τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένας ε, τεράστιος δυνάμει κίνδυνος. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή να κάνει ό,τι μπορεί για να υποχρεώσει την Λευκορωσία να σεβαστεί του, τις διεθνείς δεσμεύσεις της και, τις διεθνείς, ε, και τα διεθνή πρότυπα προβλέπει η Επιτροπή να κάνει κάτι τέτοιο, να εξασφαλίσει τους τυχόν, τυχόν κινδύνους από μια καταστροφή. Μετά από πολλές διαπραγματεύσεις φτάνουμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας γιατί το 2017 και 2018 είχαμε να αντιμετωπίσουμε πυρκαγιές και αποψήλωση των δασών. Ε, θα πρέπει να είναι σε εθελούσια βάση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συντονίζει τις προσπάθειες όταν μία χώρα ζητά αρρωγή. Αυτό θα γίνει για να μπορέσουμε να ε, διαχειριστούμε καλύτερα και τα μέσα πολιτικής προστασίας. Το RESC-EU, αυτό το αποθεματικό, θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν επαρκή σπόρους και έτσι τα ενδιαφερόμενα κράτη θα έχουν τη δυνατότητα και χρήσης αεροσκαφών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές. Αυτό αφορά και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ωραία. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση. Ο κύριος Στυλιανίδης έχει το λόγο για να απαντήσει και μετά η κυρία Γκαρντίνη. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, πριν από δύο χρόνια ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, ειλικρινά υπήρχε μεγάλη προθυμία από πολλά από τα κράτη-μέλη. Και λοιπόν ήξερα ότι είναι πιο σημαντικό να αυξήσουμε το δυναμικό μας καθώς και τους πόρους για την προσπάθεια αυτή. Καθώς και το ότι να έχουμε ένα καλύτερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση των καταστροφών και αυτό είναι σημαντικό, αλλά για μένα και όπως καταλαβαίνω και για σας, το πιο σημαντικό είναι αυτά που επέτυχε συγκεκριμένα το εξής που επέτυχε το Rescue Ενισχύουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Την κάνουμε πιο αποτελεσματική και πιο απτή. Πολύ πιο κοντά στους συμπολίτες μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και ιδιαίτερα στην παρούσα συγκυρία. Τώρα που το κοινό ευρωπαϊκή μας ε, εγχείρημα αμφισβητείται από πολλούς, δυστυχώς. Και ιδιαίτερα επειδή επίκυνται οι πολύ σημαντικέ ευρωεκλογέ. Αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε αποτελέσματα επί των υποσχέσεών μας να κατασκευάσουμε, να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που προστατεύει, που σώζει ζωές. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και σας ευχαριστώ και πάλι γι' αυτό. Αλλά μια συμβουλή να σας δώσω. Γιατί συνέλεξα πολύ εμπειρία μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια. Είναι ένα μεγάλο βήμα, αλλά ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Πρέπει να συνεχίσουμε για να αναβαθμίσουμε το μηχανισμό αυτό και σε άλλους τομείς. Ιδιαίτερα στον ιατρικό. Αυτό θα είναι ένα επόμενο ορόσημο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Στυλιανίδη. Η κύρια Γκαντίνη, συγγείται, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ χαρά τις παρεμβάσεις όλων των συναδέλφων και την επιβεβαίωση μιας ενότητας θέσεων και διάθεση συνεργασίας από όλες τις πολιτικές ομάδες, όλους τους βουλευτές, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτόμουν και το δρόμο που διανύσαμε από την προηγούμενη θητεία όταν μπήκε η έννοια της πρόληψης μέχρι σήμερα που είναι αναπόσπαστο για να μην πω προτεραιότητα κομμάτι προτεραιότητα στην πολιτική προστασία. Ευχαριστώ τον Επίτροπο που θύμισε τις δυσκολίες να πείσουμε κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχει και μία πολιτισμική σεμνότητα να αποδεχθούμε την ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια. Θυμάμαι το δίδαγμα που μάθαμε όταν η Ιαπωνία βρέθηκε μπροστά στην καταστροφή της Φουκουσίμα. Η χώρα που θεωρούσαμε η πιο προπασκευασμένη στον κόσμο δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτή την τεράστια καταστροφή. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η σεμνότητα. Η Ευρώπη που προστατεύει που παρακολουθεί είναι μια πραγματικότητα ολοένα και εντονότερη και χάρη στην προσπάθεια του Επιτρόπου και την δουλειά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουμε ένα εργαλείο που καθιστά την Ευρώπη ασφαλέστερη. Χαίρομαι που υπήρξε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τη μεταβατική περίοδο που θα μας επιτρέψει να είμαστε έτοιμοι πριν το επόμενο καλοκαίρι γιατί είδαμε ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές αυτές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό απολειών ανθρώπινων ζώων γίνονται πραγματικά το καλοκαίρι με τις δασοπυρκαγιές. Ευχαριστώ επίσης ε, και ξανά όλους σας και αφού αφιέρωσα στον Ζαμπερλέτη αυτή τη μέρα θέλω να σκεφτώ τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που σε όλη την Ευρώπη δουλεύουν για την ασφάλεια όλων μας. Στην πολιτική προστασία, στην πυροσβεστική, στους πάμπολους εθελοντές που σε πολλές χώρες δουλεύουν για μας. Η πολιτική προστασία έχει πολλές μορφές και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορέσαμε να δώσουμε τον ορισμό της πολιτικής προστασίας στην προηγούμενη θητεία. Η ενότητα ωστόσο προθέσεων και αισθημάτων είναι ένα σημαντικό τούβλο για να χτίσουμε την Ευρώπη που αγαπάμε. Μια Ευρώπη που προστατεύει, που έχει μεγαλύτερη λεγγύη και, και βοηθά τους πολίτες σας. Τους πολίτες. Ευχαριστώ όλους για την δουλειά σας. Ευχαριστούμε κύριε Γκαρντίνη. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι ασχολήθηκαν με το φάκελο αυτό και στην εισηγήτρια. Προχωρούμε στην εξέταση της έκθεσης Γκούτελαντ για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Η κυρία Γκούτελαντ δεν είναι εδώ σήμερα. Θα ακούσουμε στη θέση της την κυρία Ντάλι. Μίριαμ, παρακαλώ. Ehm, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τη Γιούτε Φίτελαντ για τη δουλειά που έκανε για την έκθεση αυτή. Όπως είπατε, ε, δυστυχώς δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα, αλλά θέλω να αποτίσω φοροτιμή στην τεράστια δουλειά που έκανε μαζί με τους συναδέλφους Κιώδης για το θέμα αυτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ πιστεύω, είμαι πεπισμένη, ότι η έντονη χρήση παραστοκτώνων στην Ευρώπη δεν είναι πλέον ε, βιώσιμη. Και η μη βιώσιμη χρήση αυτών των φαρμάκων δημιουργεί προβλήματα για το περιβάλλον, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Και μπορεί να έχει σοβαρή επίπτωση και στους γεωργούς που τα χρησιμοποιούν και στους καταναλωτές που μπορεί να έρθει σε επαφή με επικίνδυνες ουσίες που βρίσκονται στα παραστοκτόνα, στα πάρκα και στις αυλές των σχολείων. Η, βιώσιμη, η οδηγία για τη βιώσιμη χρήση παραστοκτόνων μπορεί να βοηθήσει ούτω ώστε να έχουμε μια βιώσιμη χρήση των παραστοκτόνων. Αλλά είναι σαφές, σαφέστατο ότι τα κράτη-μέλη δεν την εφαρμόζουν σωστά τι βλέπουμε. Η χρήση των παραστοκτώνων στην Ευρώπη αυξάνεται συνεχώς από τη δεκαετία του 90 και τώρα. Και παρά το ότι έχει αυξηθεί η συνειδητοποίηση για τη βιώσιμη γεωργία και παρά το ότι έχουμε καλύτερα παραστοκτώνα τώρα, τα πιο βαριά συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Υπήρξε μια κάποια πρόοδος γίνονται περισσότερος ε, έλεγχος για, την, ε, για τα ψεκαστικά μηχανήματα και ε, περισσότερη κατάρτιση για το πώς πρέπει να γίνεται αυτός ο ψεκασμός δεν έχει γίνει επαρκή για επαρκή πράγματα για την χρήση των εναλλακτικών αυτών προϊόντων. Πρέπει να υπάρχουν ποσοτικοί στόχοι τα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα σχέδια για τη χρήση των παραστοκτώνων δεν καθορίζουν πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι τους. Θεωρούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος και στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ε, ε, παρασίτων. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν σοβαρά αυτό το θέμα, γιατί οι συμπολίτε μας ανησυχούν όλο και περισσότερο και θέλουν να μειωθεί η εξάρτησή τους από τα παραστοκτόνα. Οι γεωργοί έχουν κάθε δικαίωμα να μπορούν να χρησιμοποιούν ε, ουσίες και τεχνικές που δεν θέτουν εν κινδύνο την ίδια την υγεία τους και δεν ε, έχουν τόσο αρνητική επίπτωση στο περιβάλλον και στην καλλιεργή γη τους. Χρειαζόμαστε κίνητρα που να μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση, που να βοηθήσουν τους ε, γεωργούς να μειώσουν τη χρήση αυτών των παρασιτοκτόνων και να χρησιμοποιούν περισσότερο εναλλακτικέ λύσεις ε, που να είναι πιο βιώσιμες και που δεν θα ε, εμπλέκουν ε, τη χρήση παραστοκτώνων. Η ομάδα μας θέλει να βοηθήσει όλη αυτή την προσπάθεια. Πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε άοκνα για να δημιουργήσουμε μη τοξικά περιβάλλοντα, ούτως ώστε η δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα προφυλάσσονται πλήρω από τη σημερινή ευρεία χρήση παρασυτοκτόνων. Έχουμε τα εργαλεία, πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να κάνουν την αναγκαία προσπάθεια, ώστε όλοι μας και το περιβάλλον να αποφεληθούμε από τις ισχύουσες και υπάρχουσες ε, εναλλακτικές καλύτερες λύσεις. Εάν υπάρξει καλύτερη εφαρμογή αυτής της οδηγίας, θα βοηθήσουμε πολύ ούτω ώστε να επέλθει αυτή η αλλαγή. Τέλος, υπήρξε πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των ε, σκιωδών και από πλευρά τη Γιούτα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους από τις διάφορες πολιτικές ομάδες για την επικοδομητική του στάση και την πολύτιμη στήριξή της στην εργασία της τα αργότερα Σήμερα εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα προς όλα τα κράτη-μέλη ότι στηρίζουμε όλους τους πολίτες της Ένωσης και αναμένουμε οι, τα κράτη-μέλη μας να αυξήσουν τις προσπάθειές τους για να συμβάλλουμε στην πιο βιώσιμη χρήση των παραστοκτώνων παντού στην Ευρώπη και σε ευχαριστώ πολύ. Ο, ο κύριος Ριμπέιδο για την Επιτροπή Γεωργίας. Ε, ένα λεπτό. Η κύριε Ριμπέιδο. Προαπαιτείται μια σοβαρή συζήτηση και καθόλου δημαγωγική για να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται σωστή χρήση των φυτοφαρμάκων και οι αγρότες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και το στο συμφέρον να έχουν καλλιεργήσιμες γιές με έναν υγιή υδροφόρο ορίζοντα. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι τα φυτοφάρμακα τα χρησιμοποιούν επαγγελματίας. Υπάρχουν πολλές μάστιγες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν θα πρέπει να καταργήσουμε τα φυτοφάρμακα, αλλά να είμαστε σίγουροι ποιες είναι οι δραστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται. Θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα τροφίμων το οποίο να είναι σίγουρο και βλέπουμε ότι το 97% των τροφίμων έχει υπολοιματικά στοιχεία φυτοφαρμάκων. Θα πρέπει επίσης να συγκρίνουμε τα βιολογικά προϊόντα για να δούμε ποια είναι η σύστασή τους. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Επίτροπος Κάιτης, τον οποίο και χαιρετίζω. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη, χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα στην Ολομέλεια για να συζητήσουμε την ε, βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας που συντάξατε. Θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε κοινέ ανησυχίες και κοινούς στόχους για να προστατεύσουμε τους πολίτες καθώς και την υγεία των ζώων γιατί οι Ευρωπαίοι ασχολούνται όλο ένα και περισσότερο με ζητήματα διατροφής και παραγωγής τροφίμων. Αυτό θα πρέπει να γίνεται κατά βιώσιμο τρόπο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε ένα συνεκτικό πακέτο που ρυθμίζει τα προϊόντα και τα είδη διατροφής. Η δραστική ουσία, οι δραστικές ουσίες των ε, προϊόντων θα πρέπει να εγκρίνονται από μια ευρωπαϊκή αρχή και τα φυτοφάρμακα να εγκρίνονται και σε εθνικό αλλά και κοινοτικό επίπεδο, έτσι ώστε τα προϊόντα αυτά να είναι ασφαλή για τους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον. Όπως ορίζει και η έκθεσή σας, οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν περισσότερα. Γι' αυτό η βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν εθνικά προγράμματα δράσης με στόχους, μέτρα, ποσοτικά και ποιοτικά, έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Εμείς έχουμε αξιολογήσει αυτό το πλαίσιο και έχουμε αποστείλει, είχαμε αποστείλει το 17 μία έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα εθνικά προγράμματα δράσης αποτελούν ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Υπάρχουν όμως και πολλά χάσματα, όπως προείπαμε. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν την ποιότητα των τροφίμων και θα πρέπει να ορίσουν μετρήσιμους στόχους και δείκτες για την μακροχρόνια στρατηγική μείωση κινδύνου από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Επίσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση φυτοφαρμάκων και αυτό είναι ο ακρογωνιαίος μας λήθος, τα κράτη-μέλη δεν έχουν ορίσει συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δεν θα σταματήσω να ζητώ όλο ένα και περισσότερα από τα κράτη-μέλη. Οι υπηρεσίες μου θα συνδράμουν γι' αυτό. Μετά την αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων δράσης, οι υπηρεσίες μου θα ορίσουν τις αδυναμίες αυτών των σχεδίων έτσι να ώστε να ληφθεί υπόψη στην αναθεώρησή τους. Επίσης έχουν γίνει έλεγχοι στα κράτη-μέλη για να ε, αναγνωρίσουμε εάν πραγματικά εφαρμόζεται η οδηγία. Πρόκειται για ένα μέσο για να μπορέσουμε να δούμε κατά πόσο υπάρχουν καλές πρακτικές στα κράτη-μέλη, να γίνεται ανταλλαγή επ' αυτών και αν δεν εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει περαιτέρω. Τα τελευταία, στους τελευταίους μήνες τα κράτη-μέλη ζήτησαν από την Επιτροπή να φτάσει σε εναρμονισμένους δείκτες κινδύνου. Αυτό σχετίζεται με την προστασία των προϊόντων και τώρα το Συμβούλιο αναλύει την κατάσταση, καθώς και εσείς. Θα ήθελα να δείτε θετικά αυτούς τους δείκτες που πιστεύω ότι θα δημοσιευτούν μέχρι τα τέλη του 19. Δεν είναι βέβαια το τέλος της διαδικασίας η θέσπιση αυτών των δικτών. Απλώς θα μπορέσουμε να ορίζουμε καλύτερα τους κινδύνους για την προστασία των ε, φυτών και των προϊόντων. Αυτό είναι και ο ακρογωνιαίος μας λίθος. Τα κράτη-μέλη σήμερα ε, δεν έχουν ολοκληρωμένα μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτιμούν τη συμμόρφωση ως προς την αποτίμηση κινδύνων. Το Μάιο θα οργανώσουμε ένα εργαστήριο για να ορίσουμε μία εργαλειοθήκη για την εφαρμογή αυτών των μέτρων από τα κράτη-μέλη. Η έκθεσή σας μιλά και για ουσίες χαμηλού κινδύνου